Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να σα καλέσω να καθίσετε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και θα έρθει και ο πρόεδρο Ταγιάννη, ο οποίο θα μα απευθυνθεί. Στι 5 παρατέταρτο προβλέπετε. Εν τω μεταξύ, να σας συστηθώ. Λέγομαι Αντίνα Βαλεάν. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου να προεδρεύω στο πάνελ αυτό με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τους συναδέλφους, ε, μέλη του Κοινοβουλίου και εμπειρογνώμονες. Ο τίτλος ε, του πάνελ είναι «Η επίτευξη υγιών καθαρών θαλασσών και ωκεανών». Θα ακούσουμε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις μου και κατόπιν ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Κοινοτομία θα μας απευθυνθεί, ο Ζων Ερικ Πακέ, κατόπιν θα ακούσουμε την Ιωάννα Ντρέικ, ε, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα τελευταία έτη στο να διατηρήσουν την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και κατόπιν θα ολοκληρώσουμε με ομιλητές από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Δυστυχώ δεν θα έχουμε πολύ χρόνο για διάλογο. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας δύο λόγια. Δυναμή του δικού μου ρόλου. Ξέρουμε ότι οι ωκεανοί αποτελούν το 7% της επιφάνειας του πλανήτη και το 97% του είδους καλύπτει πάνω από το 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ε, θάλασσα μας δίνει κινητικότητα, ψυχαγωγία, φάρμακα, αλλά επίσης οι ωκεανοί ρυθμίζουν το κλίμα, μας ε, δίνουν οξυγόνο και απορροφούν μεγάλο ποσοστό των εκπομπών του διεξιδίου του άνθρακα. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες που προφέρονται από τους ωκεανούς είναι ζωτική σημασίας για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Οι, ανθρωπινές, ε, οι δραστηριότητες έχουν ε, μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στο οικοσυστήμα των ωκεανών λόγω της κλιματικής αλλαγής, της οξύνησης, της υπερελίευσης, της ρήπανσης και των σκουπιδιών, της καταστροφής, των οικοτόπων και των χωροκακτητικών ειδών. Όλα αυτά έχουν καλυφθεί από νομοθεσία και από έγγραφα με κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε αναλάβει δράση προκειμένου να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας των νομοθετημάτων. Οι συνάδελφοι στη συνέχεια θα σας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχει συμπεριλάβει το Κοινοβούλιο στην νομοθεσία προκειμένου να βελτιώσει το καθεστώς των ωκεανών. Όμως η θέση σε ισχύ της νομοθεσίας αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Σε ό,τι αφορά τις γενικές πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική πριν 11 χρόνια έθεσε τον στόχο κλειδί να διασφαλίσει ένα καλό περιβαλλοντικό καθεστώς ε, όλων των ε, θαλάσσιων υδάτων μέχρι το 2020. Σε επίπεδο ε, Ηνωμένων Εθνών, ο στόχος βιώσιμη ανάπτυξη 14, δηλαδή να χρησιμοποιούνται οι ωκεανοί και θάλασσε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει τεθεί στην, στο θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το να μπορούμε να πετύχουμε του στόχου αυτού ε, έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μα Πέρσι, η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για την εξολόγηση προγραμμάτων των κρατών μελών για τα μέτρα που είχαν πάρει δυνάμει τη οδηγία ε, πλαίσιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχαν καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν ε, τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, η εξολόγηση δείχνει ότι όλες οι πιέσει στο περιβάλλον στο θελάσσιο περιβάλλον δεν καλύπτονται κατάλληλα από τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Τα ίδια τα προγράμματα έχουν ε, ψηλά ποσοστά φιλοδεξίας ε, να πετύχουμε ένα καλό περιβαλλοντικό καθεστώς μέχρι το 2020. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το 2017 πολλές πολιτικές ε, ε, είχαν τεθεί σε εφαρμογή και παρά αυτό το γεγονός, παρά δηλαδή το ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσματα, οι πιέσεις ε, στο θαλάσσια περιβάλλοντα συνεχίσουν να αυξάνονται. Πράγματι, η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2015 ε, της ε, περιβαλλοντικής στρατηγικής μας έδειξε ότι έχουν γίνει πολλές ε, προσπάθειες αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σε κάποιους τομείς δείχνει ότι συνεισφέρει στο στόχο 14 το SDG, δηλαδή έχει δεσπίσει προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τα ε, θαλάσσια απόβλητα. Είχαμε το 1998 την πρώτη σχετική νομοθεσία. Από τότε η ρήπανση με πλαστικά των ωκεανών έχει διαβλάβει τέτοιο μέγεθος και θεωρείται ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε περισσότερο πλαστικό από ψάρια στους ωκεανούς. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ευρεία σειρά εργαλείων όπως ε, περνούντος χάρη ε, κανονισμούς ε, για την συλλογή των αποβλήτων και τον οδηγία για τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων στους λιμένες. Και αφού έχουμε συνεισφέρει στην υιοθέτηση του πακέτου για τα απόβλητα το 2018 που θα αυξήσει τους στόχους ανακύκλωσης, και πρόσφατα, ε, τον προηγούμενο Δεκέμβριο, θετήσαμε για την οδηγία για τα πλαστικά μία χρήση. Εκεί θέτουμε πιο αυστηρούς κανόνες για τα πλαστικά προϊόντα και τη συσκευασία μεταξύ που είναι μεταξύ των 10 ε, πρώτων προϊόντων που βρίσκουμε στις παραλίες. Η οδηγία θα απαγορεύσει ε, τη χρήση κάποιων πλαστικών μιας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικέ και συγκεκριμένα μέτρα θα εισαχθούν για να μειωθεί η χρήση των ε, υλικών ε, πλαστικών προϊόντων ε, που απορρίπτονται και για τα οποία δεν υπάρχουν εναλλακτικέ. Είναι λοιπόν σαφέ ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και φροντίδα οικιανή και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με ισχυρή διεθνή συνεργασία. Υποστηρίζουμε πλήρω την ανάπτυξη νομικών δεσμευτικών μέσων όπως η βιώσιμη χρήση και η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας δυνάμει της Η μείωση της ανθρώπινης πίεσης στους ωκεανούς είναι μια δέσμευση που θα πρέπει να αναλυφθεί σε όλα τα επίπεδα από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τον μεμονωμένο καταναλωτή. Και με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζάνερικ Πακέ, τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και καινοτομία. Παρακαλώ. Κύριε Πακέ, έχετε πέντε λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτό το πάνελ. Και εφόσον μίλησε ήδη ο Επίτροπος, λίγα λόγια για το πού βρισκόμαστε στην έρευνα σχετικά με τους ωκεανούς. Κοιτάζουμε το μέλλον και την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος πλαισίου για τον ορίζοντα της Ευρώπης. Αυτό υπόθηκε και στην προηγούμενη σύνοδο και θα το ακούτε και από όλα τα μέλη του πάνελ. Οι ωκεανοί μεταβάλλονται ε, ε, εκ βάθρων από όλε τις απόψεις. Κυρίως από την άποψη τη μετεωρολογική. Ε, οι νέε κανονικέ συνθήκε είναι το απρόσμενο των αλλαγών του καιρού. Οι καταιγίδε ε, διαρκώ είναι διαφορετικέ. Είδατε ότι ο τυφώνα στη Μοζαμβίκη είναι ένα περιστατικό που δεν θα είχε λάβει χώρα ούτω υπό άλλε συνθήκε. Και βεβαίω ο καιρό επηρεάζει και το τι γίνεται στου ωκεανού. Το θέμα του οξυγόνου στου ωκεανού. Οι ωκεανοί ε, παράγουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και αυτό όμω αλλάζει. Οι ωκεανοί παράγουν τα τρόφιμα που καταναλώνουμε αλλά και εκεί επισυμβαίνουν αλλαγέ, Οι ωκεανοί είναι η μεγαλύτερη αποθήκη, η δεξαμενή άνθρακα που διαθέτουμε. Επίσης, η σχέση των ωκεανών σε σχέση με το λιώσιμο των πάγων ε, μεταβάλλεται, ε, αλλάζει η στάθμη της θάλασσας και ο ρυθμός ανόδου της και εκεί θα συνεχιστούν οι αλλαγέ, αλλά τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ήδη το 2016 το μέσο επίπεδο της θάλασσας ήταν 20 εκατοστά παραπάνω από ό,τι πριν από έναν αιώνα. Και με τις τωρινές τάσεις υπολογίζουμε 60 εκατοστά συνολικά παραπάνω μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτή τη στιγμή η ωκεανή είναι η ισχυρότερη πηγή βιοπικιλότητας. Αυτό είναι γνωστό για τον πλανήτη μας και το γονιδιωμά του, αλλά αυτό μεταβάλλεται γοργά. Οι ωκεανή όμως είναι και το νέο σύνορο που αν ξεπεράσουμε θα μετρήσουμε κατά πόσο αν είμαστε καινοτόμοι. Υπάρχει το θέμα της γαλάζιας οικονομίας που μπορεί να φτιαχτεί με βάση τους ωκεανούς μας. Ενέργεια, υλικά, ε, ηχθειοκαλλιέργεια και βιολογικά προϊόντα, όλα αυτά είναι στοιχεία που έχουν σχέση με τους ωκεανούς και θα μπορέσουν να ενισχύσουν και την οικονομική μας πρόοδο. Εάν όμως μεταβαλλόνται τόσο ε, βαθιά οι ωκεανοί και είναι τόσο σημαντικοί για το μέλλον μας, ξέρουμε αρκετά καταλαβαίνουμε αρκετά άραγε για τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Ε, εδώ ακούσαμε να λένε όλοι οι μελτές ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι το 2030 έχουμε μία δεκαετία για τους ωκεανούς, για να αφοσιωθούμε στο θέμα των ωκεανών, να τους καταλάβουμε, να τους μελετήσουμε και να βρούμε λύσεις. Το παράδοξο όμως είναι ότι Ξέρουμε πολύ περισσότερα για το ηλιακό μα σύστημα και το διάστημα από ό,τι για του ωκεανού. Οι ωκεανοί πρέπει να χαρτογραφηθούν πλήρω και δεν γίνονται αρκετά προ στιγμή ε, ούτε διεθνώ ούτε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν το Horizon Europe, θέτοντα ω στρατηγικό τομέα ε, του ωκεανού στι προτεραιότητε του προγράμματο, θα βοηθήσει για του στόχου των φυσικών πόρων. Δεν μπορούν ε, βεβαίω τα ευρωπαϊκά προγράμματα να αντιμετωπίσουν ε, όλε αυτέ τι ανάγκε μόνα του. Χρειάζονται συνδυασμένε προσπάθειε, αλλά ήδη αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα η ανάγκη ευρωπαϊκή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ασχοληθούν με αποστολές έρευνας που θα ε, αφορούν εν μέρη τους καθαρούς ωκεανού και θάλασσες. Και αυτέ οι αποστολές θα αλλάξουν εντελώ τα δεδομένα. Διότι όχι μόνο θα επιστήσουν την προσοχή των συμπολιτών μας στο θέμα των ωκεανών, αλλά θα αποσχολήσουν και τις ευρωπαϊκές ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει τι γραμμή πλεύσης θα ακολουθήσει εμείς, τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τι απαντήσεις θα δώσουμε στα προβλήματα των ωκεανών. Να μένονται λοιπόν από εμά πολύ συγκεκριμένε προτάσει ε, για να πετύχουμε τα αποτελέσματα και με λύσει που θα εφαρμοστούν για να είναι χειροπιαστά τα αποτελέσματα. Η πρώτη φάση ξεκίνησε. Η πρώτη αποστολή έχει μια επιστημονική ατζέντα, όχι μόνο και ερευνητική ατζέντα, όχι μόνο βάσει του Horizon 2020, γιατί εκεί θέλουμε να συντονίσουμε τις προσπάθειες μεταξύ κρατών μελών σε όλη την Ευρώπη και με δημόσιες και ιδιωτικές ε, συνεργασίες, αλλά χρειάζεται όλοι οι φορείς να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια βαθιά αλλαγή, πραγματική αλλαγή, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την ατζέντα, αυτόν τον κατάλογο προτεραιοτήτων, με την πολιτική για του ωκεανού, όπω είπε και η κυρία Βαλιά. Διότι δεν μπορεί η έρευνα μόνη τη να αλλάξει τα πράγματα στην πράξη, αλλά η χάραξη πολιτική βάσει των γνώσεων που η έρευνα έχει προηγουμένω προσφέρει και των λύσεων που μπορεί να προτείνει. Αυτά θα κάνουν την πραγματική διαφορά. Να διασυνδέσουμε την έρευνα και την επιστήμη με τι ε, πολιτικέ προτεραιότητε. Αυτό είναι η ουσία. Και αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι ωκεανοί μα και εκεί όπου υπάρχει και συγχρηματοδότηση. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε για του ωκεανού ε, στην μελέτη τη μελλοντική χρηματοδότηση του Horizon 2020. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διαπραγματεύσεων για το Horizon 2020. Θα ολοκληρωθεί μάλλον τι επόμενε ώρε η σχετική διαπραγμάτευση για το Horizon 2020. Και όσοι ε, ενδιαφέρονται για το θέμα των ωκεανών, α ενώσουν τι δυνάμει του για να συζητήσουν τι προτεραιότητε του ορίζοντα 2020 για την ερχόμενη χρονιά. Οπότε όταν αρχίσει να τρέχει στι αρχέ του 2021 το πρόγραμμα αυτό, να ξέρουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε και πρέπει να κάνουμε για αυτέ. Η Ευρώπη είναι ναυτική, είναι θαλάσσια. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτή παγκοσμίω, 68.000 χιλιόμετρα. Δυο φορέ περισσότερα από τη Ρωσία και τρει από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, έχουμε τον πολιτισμό και την κουλτούρα μα να βασίζονται στου ωκεανού. Είμαστε μια ένωση ωκεανών. Και εδώ τα προγράμματά μα θα πρέπει να συνδυαστούν με φιλοδοξότερε κρατικέ και δημόσιε πολιτικέ. Οι ωκεανοί βρίσκονται στην καρδιά του περιβαλλοντό μα. Ευχαριστώ. Okay, okay, understood. Um, okay, thank you. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πακή. To Madam Drake. Και με χαρά θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τζέικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλεάν για την ευκαιρία που μου δίνετε ο πλανήτης μας καλύπτεται κυρίως από τη θάλασσα. Ε, άρα ε, η καλή κατάσταση των θαλασσών είναι απαραίτητη για την ίδια τη ζωή ε, στη γη. Το είπαν πολλοί προαλήσαντες και ο Ζαν τώρα μόλις. Σήμερα όμως έχουμε έρθει εδώ για να αποτυπώσουμε ε, την κατάσταση, τι έχουμε κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίσουμε πού βρισκόμαστε και τι απομένει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Η θάλασσα πάνω απ' όλα είναι η πηγή ε, πολλών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που παράγουν υπηρεσίες και ε, αποφέρουν πόρους από τους οποίους τόσο πολύ σήμερα εξαρτώμαστε. Ωστόσο αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες είτε είναι αλληλεία, ναυτιλία, γεωργία, ενέργεια και πολλές ακόμα ασκούν πιέσεις στη θαλάσσια ζωή, στους οικοτόπους και απειλούν πολλές φορές την πρωταρχική ε, λειτουργία των ωκεανών μας, που είναι να διαφυλάξουν και να διατηρήσουν ζωντανό τον ίδιο τον πλανήτη μας. Πολύ συχνά ε, είμαστε πολύ φιλόδοξοι, έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και σεμνινόμαστε γι' αυτό, γιατί όντως πρέπει να είναι καθολικό, προστατευτικό και να μπορεί να εφαρμόζεται. Όλοι αυτοί είναι στόχοι ένα πλαίσιο για την αλία, για το περιβάλλον ε, και ε, ε, καθώς επίσης με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις όλα αυτά συνδέονται και συνδυάζονται. Μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά χάρη σε αυτό το πλαίσιο ενωμένα τα κράτη-μέλη προοδευτικά κάνουν κάποιες βελτιώσεις έτσι ώστε να φτάσουμε στους στόχους. Βήματα για να είμαστε πιο συντονισμένοι και με στρατηγική να προστατεύουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Ας πούμε, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να έχουν μια καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, δηλαδή μέχρι το 2020 θάλασσες καθαρές, παραγωγικές και υγιείς. Ε, αν δούμε όμως τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος, αν αποτυπώσουμε την κατάσταση, απομένουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν. Και είναι μάλλον απίθανο να είναι σε καλή κατάσταση το περιβάλλον ε, ε, παντού και πουθενά ε, και, και για όλα αυτά τα θέματα μέχρι το 2020. Αυτό επίσης αντανακλά τη συνολική εικόνα των ωκεανών που βρίσκονται σε ανισχυτική κατάσταση. Ε, βέβαια όλα είναι προβλήματα εφαρμογής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τόνισε αυτό επανειλημμένα σε διάφορες εκθέσεις. Ε, αυτό όμως οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Και οι άλλοι παράγοντες ποιοι είναι, για παράδειγμα. Χρειάζεται περισσότερη καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε αποτελέσματα επιτόπου. Επιτρέψτε μου εδώ να σας αναφέρω το παράδειγμα των πλαστικών μιας χρήσης. Προηγήθηκε το πρώτο πάνελ που αναφέρθηκε στη διακυβέρνηση, που και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Δεν θα επιμείνω τώρα σε αυτό. Η περιφερειακή συνεργασία είναι βεβαίω κομβική σημασία για ε, την επιρροή μα στη θάλασσα, όπω είναι η απώλεια τη βιοπικιλότητα, η ρήπανση και η απώλεια της βιοπικιλότητας είναι αχαλήνοτη. Εμείς έχουμε εισβάλλει στη θαλάσσια ζωή με τις δικές μας δραστηριότητες, υποβαθμίζουμε το πολύτιμο οικοσύστημα και τους οικοτόπους, αλλά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ε, τα οικοσυστήματα και να ε, βοηθήσουμε ε, να ανακτώνται τα είδη και να αναπαράγονται αν δεν ορίσουμε προστατευόμενες περιοχές για τη θαλάσσια ζωή. Άσυλα. Ε, χάρη στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των θαλασσών, τώρα έχουμε περίπου, περίπου 11% των θαλασσών να καλύπτονται, ενώ παγκοσμίω αυτό το ποσοστό είναι στο 7%. Χρειαζόμαστε όμως μια ε, γερή όθηση για να γίνεται σωστή διαχείριση με σωστά μέτρα συντήρησης και διαχειριστικά σχέδια έτσι ώστε να έχουμε και οικολογικά ωφέλη και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη απορρίμματα, τα απόβλητα στη θάλασσα είναι σύμβολο της ε, αναπαραγωγικής και αναποτελεσματικής μας οικονομίας. Τα ρίχνουμε στη θάλασσα και στις ακτές τα σκουπίδια αντί να τα ανακυκλώνουμε και να τα επαναχρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια βάση ε, στους λιμένες για την καταπολέμηση της ρήπανσης των θαλασσών από πλαστικά. Ωστόσο, ε, επίκυνται και άλλες προσπάθειες υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν γενικά την οικονομία και την ε, ποιότητα της ε, ανακύκλωσης των πλαστικών. Έχουμε νομοθεσία για την ε, μία χρήση για αλευτικά εργαλεία που χάνονται στη θάλασσα και επίσης έχουμε βελτιωμένους κανόνες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων. Γνωρίζουμε όμως αρκετά για τη θάλασσα, τα είπε ο Ζαν Ερίκ προηγουμένως. Προφανώς υπάρχουν κενά γνώσεις που θα πρέπει να καλύψουμε και εδώ ε, αυτό αφορά την αλία, τα ίδια τα απόβλητα στη θάλασσα, το θόρυβο στο βυθό, τον υποβρύχιο θόρυβο και ε, ε, την καινοτομία ε, και τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα και για τις υδατοκαλλιέργειες. Τέλος, είναι ε, σίγουρα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι γίνονται τόσο πολλά για τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Επίσης, μπορούν ακόμα να γίνουν πολύ περισσότερα και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από κοινού, φωτίζουμε αυτή την πτυχή τις απειλές και τις ευκαιρίες θα πρέπει από κοινού να δούμε πώς θα προστατεύουμε τους ωκεανούς, πώς θα δρούμε, πώς θα δρέπουμε τους καρπούς όλοι και πώς θα σεβόμαστε τους ωκεανούς γιατί πραγματικά αξίζουν τόσο πολύ το σεβασμό μας. Thank Ευχαριστώ πολύ και τώρα με χαρά ανακοινώνω ότι θα πάρει το λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος Αντώνιο Ταγιάννη. Ζητώ συγγνώμη. Θα πρέπει να κατέβουμε στην πρώτη σειρά των εδρών και θα επανέλθουμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώ ήρθατε στο ημικύκλιο του Ευρωκοινοβουλίου. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Κιασίνε Μέσνερ, ειδική επιτετραμένη του Ευρωκοινοβουλίου μας για τις θαλάσσιε υποθέσει. Βρίσκεστε στην καρδιά της διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση και είστε και ο διευθυνονούς, ο κύριο Βέλα, ο κύριο Μουέδας, ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, ο κ. Καντέκ, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Αλία, η κ. Βάλεαν, εκπρόσωπο τη Επιτροπή ΕΜΒΗ, ο κ. Χένκελ, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ήτρε. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να υποδεχόμαστε στο υποκύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω από χίλιε πολίτε, ερευνητέ, επιστήμονε, πολιτικού ηθήνοντε, επιχειρηματίε και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και των ενώσεών τη. Στην αρχή τη θητεία μα διοργανώσαμε 11 ε, συνόδου διασκέψει υψηλού επίπεδου μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτιστική κληρονομιά, την Αφρική, την ε, ψηφιακή η διάσταση, τη μετανάστευση και το καθεξής. Ήρθαν πολίτες, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, ενώσει, φορείς για θέματα που είναι κέρια σημασία για την Ευρώπη και τους πολίτες μας. Σήμερα θελήσαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα ύψης της σημασίας. Το μέλλον των ωκεανών μας. Πρόκειται για μια ε, σύνοδο που θελήσαμε με μεγάλη αποφασιστικότητα να διοργανώσουμε και ευχαριστώ και την ε, δική μου ε, υπετετραμένη την κυρία Μάισνερ για την διοργάνωση και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε, λέγαμε πριν τις ευρωεκλογέ. Το συζητάγαμε διαρκώς. Ένα γεγονός τέτοια σημασίας δεν μπορούσαμε να μην επιμείνουμε στη διοργάνωσή του. Είναι για το περιβάλλον, είναι για την ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, τα πλαστικά. Είμαστε στην πρώτη γραμμή στην μπροστοφυλακή. Για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του πλανήτη μας πρέπει εμείς οι κυβερνώντες να είμαστε σε θέση να δράσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο. Η ε, διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η περιβαλλοντική της διεύθυνση πρέπει να είναι υπόδειγμα για όλους τους διεθνείς παράγοντες. Θέλουμε περισσότερες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος για να αναλάβουν την, τους, την κοινωνική τους ευθύνη, να προωθήσουν την καινοτομία, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε ένα σημαντικότατο ψήφισμα το οποίο ε, βλέπει θετικά την δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν καθαρό πλανήτη για όλου. Θέλουμε μια οικονομία σε άνθηση, σύγχρονη, ε, περιβαλλοντικά ουδέτερη. Θέλουμε την απαλλαγή από τον άνθρακα με το στόχο μηδενικών εκπομπών ε, και τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου στο 2050 παροτρύνουμε τα κατημέρια να αναλάβουν δεσμεύσει για να πετύχουν το στόχο αυτό. αναγνωρίζουμε όμω ότι υπάρχουν και κίνδυνοι από τι κλιματικέ αλλαγέ. Βάσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο μεταξύ του 2010 και 2016, οι μέγιστε απώλειε τη Ένωση λόγω των μετεωρολογικών και ακραίων καιρικών συνθήκων έφτασαν τα 12 δι ευρώ, 8. Εάν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα και με υψηλές εκπομπές, ε, το ετήσιο κόστος των πλημμυρών μπορεί να φτάσει τα χίλια δις ευρώ μέχρι το 2020 μέχρι το 2100. Μέχρι το 2030 το 50% των ακατοικούμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίσει προβλήματα λειψιδρίας. Γι' αυτό χρειάζεται μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για να συμπεριληφθούν τα περιβαλλοντικά θέματα σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ε, πολιτικής μας για το εμπόριο. Όλες οι εμπορικές μα συμφωνίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με τη Συμφωνία των Παρισίων είτε για να βελτιώσουμε τη διεθνή δράση κατά των κλιματικών αλλαγών, είτε για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν συνθήκες ε, και όροι ισοτιμία στη δράση των επιχειρηματιών μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά μα ε, διεθνώ και όλε μα προσπάθειε για το κλίμα, για την οικονομία να ενισχύονται ε, αμοιβαίω. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τι λύσει για το περιβάλλον, για την ψηφιακή μα δράση, για την καθαρή ενέργεια, να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τι μελλοντικέ δεξιότητε και να δημιουργήσουμε εκατομμύρια θέσει εργασία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε με αυτόν τον τρόπο τους ωκεανούς και να τους ρηπαίνουμε. Θα πρέπει την ευφυή χρήση των ωκεανών και την πάυση της ρηπανσής να τους θέσουμε μεταξύ των στόχων της χιλιατίας του ΟΗΕ. Είμαστε μεταξύ των πρώτων που ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Στην διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς, τον Ιούνιο πριν από δύο χρόνια, ε, μπορέσαμε να καθορίσουμε 19 σοβαρούς στόχους, φιλόδοξους στόχους, για να σταματήσει η απόρριψη από πλήτων στη θάλασσα, να παρακολουθείτε η κατάσταση των υδάτων και να προχωρήσουμε στη διακυβέρνηση των ωκεανών. Θέλουμε νομοθετικά εργαλεία διεθνούς επίπεδου ε, για την βιοπικιλότητα στη θάλασσα και την παράνομη ηλία. Θέλουμε ένα μοναδικό νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις δράσεις που έχουν σχέση με τους ωκεανούς. Σήμερα έχουμε πάνω από 150 εκατομμύρια τόνου πλαστικού στους ωκεανούς μας. Κάθε χρόνο καταλήγουν στη θάλασσα επιπλέον 8 τόνοι. 8 εκατομμύρια τόνοι. Ε, με αυτό το ρυθμό μέχρι το 2050 στι θάλασσε θα έχουμε περισσότερα πλαστικά από τη ψάρια. Είναι μια ζημιά περιβαλλοντική αλλά και οικονομική γιατί πλήττει τον τουρισμό και την ε, αλία. Το 70% των ε, αντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα, των ε, διαφόρων προϊόντων, είναι μιας χρήσης. Γι' αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση τέτοιων πλαστικών μέχρι το 2021. Αυτό ζήτησε το Κοινοβούλιο. Το πακέτο μα για την ε, κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε την περσινή χρονιά αλλάζει τον τρόπο παραγωγή μα. Θέλουμε ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή του που είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον. Εάν ανακυκλώσουμε ένα εκατομμύριο τόνων πλαστικού, θα απαλλάξουμε του δρόμου μα. Είναι μάλλον σε ένα να βγάζουμε του δρόμου μα ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα. Την, περασμένη εβδομάδα στην Αυλομέλεια του Στρασβούργου εγκρίναμε μια οδηγία που δεν θεωρεί αυτομάτω ω παραγωγό έναν αλλιέ ο οποίο ε, φέρνει και ε, εκφορτώνει απόβλητα που τυχαίω πιάστηκαν στα δίχτυα του. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε το κόστο τη αποκομιδή και δίνουμε τη δυνατότητα να μην ε, μένουν τόσα πολλά απόβλητα στι θάλασσε. Δίνουμε κίνητρο στα σκάφη να ασχολούνται με τα ίδια του τα απόβλητα και την αποκομιδή του και να τα πηγαίνουν στα λιμάνια, όπου θα δημιουργηθούν κατάλληλε εγκαταστάσει. Γι' αυτό ελπίζω τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στα δυνατόν πιο γρήγορα αυτή την οδηγία. Με περίπου 5,5 εκατομμύρια εργαζομένου, υποστηθέμενη αξία των 500 δι ευρώ ετησίω, η γαλάζια οικονομία είναι προφανώ κέρια σημασία για την Ευρώπη. Κάποιοι τομεί όμω έχουν και άλλα περιθώρια ανάπτυξη. Σήμερα το 75% του εξωτερικού μα εμπορίου και το 37% των συναλλαγών στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά γίνονται μέσω θαλάσση. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία για να έχουμε θαλάσσιε μεταφορέ που να είναι αποτελεσματικότερε. Ο νέο προπολογισμό τη Ένωση για το 2021 έω 2027 θα πρέπει να προβλέπει μέτρα υποστήριξη αυτού του σκοπού, αυτή τη στρατηγική. Οι καθαρέ θάλασσε και οι καθαρέ ακτέ θα πρέπει να είναι κριτήρια δύναμη τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, είναι ένα πόρο οικονομικού, εμπορικού και τουριστικού χαρακτήρα, μοναδικό παγκοσμίω. Σε ό,τι αφορά την μηχανή τη Αλία, αυτή προσφέρει στου Ευρωπαίου καταναλωτέ περίπου 6,5 εκατομμύρια τόνο ψαριού ετησίω και δίνει δουλειά σε 350.000 Ευρωπαίους. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον τομέα της αλίας και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Θα πρέπει <clears throat> να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην βιώσιμη αλεία. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει, σε όλη αυτή τη θητεία μάλλον, εργαστήκαμε για τον κανονισμό, για την συλλογή δεδομένων και αυτόν για, την για τον εξωτερικό μας στόλο, τον εξωενωσιακό. Ε, για να ολοκληρώσω, πολλές ευρωπαϊκές ε, ανακαλύψεις και προτάσεις και, και ε, πρωτοποριακά βήματα ήταν αποφασιστικά για την διαφύλαξη του πλανήτη. Όπω ε, τα βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα ανακυκλώσιμα υλικά και η τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών. Με το πρόγραμμα Κοπέρνικο ε, συγκεντρώσαμε θεμελιώδη στοιχεία για να καταλάβουμε καλύτερα τον πλανήτη μα και να μπορούμε να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Να γιατί η διαστημική πολιτική χρησιμεύει και για να προασπιστούμε τη φυσική μας κληρονομιά, να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να έχουμε καλή και σωστή διαφύλαξη του πλανήτη. Οι υπηρεσίες του Κοπέρνικου είναι ένα σημαντικός πόρος για την διαχείριση των αστικών περιοχών, την βιωσιμή ανάπτυξη, την προστασία της φύσης, τον περιφερειακό χωροτοξιακό σχεδιασμό, τη γεωργία, την αλία, την υγεία, την ε, προστασία των πολιτών, τις οικοδομές, την ε, μεταφορά και τον τουρισμό. Γι' αυτό ζητάμε μεγαλύτερες προσπάθειες ε, και περισσότερε επενδύσεις για καινοτομία και έρευνα. Είναι αλήθεια ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει αύξηση στο πακέτο αυτό που ήταν ορίζοντα 2020 και τώρα θα ονομάζεται ορίζοντα Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε φιλοδοξότεροι. Η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου προβλέπει κι άλλη αύξηση επιπλέον σε αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητήσαμε από το 50% να φτάσουμε στα 120 δις ευρώ και ζητήσαμε το 30% όλων των δράσεων προβλέποντα τον επόμενο προπολογισμό της Ένωσης, ε, δηλαδή το 35% του ορίζοντα Ευρώπη, να αφορά μέτρα βιωσιμότητας. Για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις οικονομίες κλίμακας και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να έχουμε κοινού πόρους στο ύψος των προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και επιμένω, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από την Ευρώπη και να λένε ότι είναι δικό μας το φταίξιμο. Τώρα πρέπει να, ε, παίξουν το, να πάρουν μέρος στο παιχνίδι αυτό και τα κράτη-μέλη. Το περιβάλλον, η έρευνα, η καινοτομία, η βιομηχανία, η βιομηχανία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένε. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι ενώσει και επιχειρήσει είναι το κλειδί για, την ε, ε, για το σωστό συνδυασμό περιβάλλοντο και καινοτόμου ανταγωνιστική ε, οικονομία. Θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι φίλη των ωκεανών. Θέλουμε να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο και από την σκοπιά τη περιβαλλοντική διπλωματία, όπω κάναμε με την COP24 στο Κατόβιτσα το Δεκέμβρη, και με συγκεκριμένε δεσμεύσει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια όλων σα. Είναι μια πρόκληση που καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε και να την κερδίσουμε μαζί, να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Ε, οι ευχαριστίε μου, οι ευχαριστίε όλου αυτού του κοινοβουλίου πηγαίνουν και κατευθύνονται προ εσά. Εσά που δώσατε αυτέ τι μάχε. Η δική μου η δέσμευση προ του συναδέλφου του κοινοβουλίου είναι ότι μπορείτε και όλων μάλλον των συναδέλφων του Κοινοβουλίου ότι μπορείτε πάντοτε να υπολογίζετε σε εμά και στην υποστήριξή μα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ας συνεχίσουμε με το δεύτερο πάνελ. Είχαμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ε, Γενική Διευθύνση για το Περιβάλλον, την κυρία Ντρέικ. Τώρα να δώσω το λόγο στου επόμενου ομιλητέ. Ε, είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ασχοληθεί με το θέμα θα ξεκινήσω με τον Μάρκ Ντεμεσμάκερ, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να περιοριστείτε στα τρία λεπτά. Αυτό απαιτεί η οργάνωση της διάσκεψης. Παρακαλώ τρία λεπτά κύριε Ντεμεσμάκερ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Στα αγγλικά, καλησπέρα σε όλους σας. MEP for ECR Group. Είμαι ευρωβουλευτής από την ομάδα ECR Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Ασχολούμουν σε αυτή τη θητεία με όλα τα θέματα της κυκλικής οικονομίας και το, τη νέα ρύθμιση για τα πλαστικά μιας χρήσης. Πολλά ε, ακούστηκαν ήδη. Το πλαστικά είναι ένα υλικό πολύτιμο και χρήσιμο και έχουν τη θέση του στην κοινωνία μας. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε πλαστικά σήμερα είναι και αφορητός αλλά και πανάκριβος. Επιπλέον, η ανακύκλωση πλαστικών και συλλογή τους παραμένει πολύ χαμηλή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 5% της αξίας των συσκευασιών, των πλαστικών συσκευασιών παραμένουν στην οικονομία μας. Άρα το 95% της αξίας χάνεται. Και είναι βασική η πρόκληση να διαχειριζόμαστε τα πλαστικά με τρόπο βιώσιμο όσο και ε, υπεύθυνο σε όλη την αλυσίδα. Η στρατηγική για τα πλαστικά θα πρέπει να είναι μοχλός για να ενθαρρύνει και να κινητροδοτεί για νέα μοντέλα, για νέες λύσεις, ε, κοινέ δεσμεύσεις και δράσεις από όλους τους ε, ενεχομένους την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία όχι απλώς να τα ξαναπούμε αλλά να προχωρήσουμε και σε δράσεις. Θα δούμε τι θα βγει από το τριμερή διάλογο και τη συμφωνία για τα πλαστικά μιας χρήσης ε, στον οποίο κατέληξαν μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο ε, που δεν θα ξεχάσω ποτέ ούτε εγώ ούτε ο Επίτροπος Βέλα. Πάντω ήταν καλό το αποτέλεσμα και είμαι πεπισμένο ότι αυτή η νομοθεσία είναι κρίσιμη για τη μετάβασή μα προ την κυκλική οικονομία, αλλά και προς ένα βήμα στο να κρατήσουμε τα απορρίμματα αυτά τα πλαστικά μακριά από τι θάλασσε τα πελάγια και του ωκεανού μα. Ιδιαίτερα τα πλαστικά απόβλητα είναι μεγάλο πρόβλημα πέρα από τα υπόλοιπα σκουπίδια για τι θάλασσε και του ωκεανού. Και όπως είπε και ο πρόεδρο, πρέπει να αποφύγουμε να καταλήγουν στη θάλασσα τελικά, ε, να έχουμε περισσότερα πλαστικά απόψα ψάρια στο μέλλον. η δέσμη ε, μιλάει για τα 10 κοινότερα ε, προϊόντα πλαστικών που βρίσκουμε στις ακτές μας στην Ευρώπη και το Κοινοβούλιο χαίρεται που θα απογορευθούν ε, τα προϊόντα ε, από ε, όξο αποσπόμενα πλαστικά. Το θέμα είναι ότι δεν, δεν ε, ε, διαλύονται αυτά, αλλά γίνονται ε, πάρα πολύ μικρά σωματίδια πλαστικού. Τα κράτη-μέλη επίση θα πρέπει να μειώσουν τους πλαστικούς περιέκτες τροφίμων και τα πλαστικά κυπελάκια μιας χρήσης, ποτήρια δηλαδή. Επίση, το κόστος καθαρισμού είναι πολύ μεγάλο και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι κάνουμε βήματα προ τα εμπρό. Έχουμε δεσμευτικό στόχο για ε, ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών ποτών μέχρι ε, το 2029 κατά 90%. Τα πλαστικά μπουκάλια ε, αναψυκτικών ποτών και τα λοιπά είναι αυτά που βρίσκουμε περισσότερο στις ακτές μας. Και καταφέραμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη μέχρι το 2030 μέχρι το 2030 να είναι το 30% ανακύκλωσιμο προϊόν στις συσκευασίες. Επίσης, τα πλαστικά φίλτρα τσιγάρων είναι το, το δεύτερο μετά τα μπουκάλια ε, που βρίσκουμε. Μέχρι 500 λίτρα νερού μπορεί να ρυπάνει μία πλαστική γόπα από τσιγάρο και θα πρέπει καπνοβιομηχανοί να τα ξέρουν αυτά και να ε, πληρώνουν το κόστος της συλλογής σε δημόσιους χώρους. Είναι σίγουρα μια πολιτική συγκυρία πάρα πολύ σημαντική, την υποστηρίζουν οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών για να περάσουμε σε μια μετάβαση, σε μια κυκλική οικονομία με ανακύκλωση πλαστικών. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε αυτές τις οδηγίες και η μετάβαση ε, στην κυκλική οικονομία θα μας κάνει να κάνουμε τις χωματερές χρυσορυχία. Και τελικά αυτή η σούπα των πλαστικών στους μπορεί να γίνει ένα τεράστιο γαλάζιο λιβάδι. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρικάρτο Σεραοσέντο, ο οποίο είναι μέλο τη Επιτροπή Αλία. Ελπίζω να μείνετε στα τρία λεπτά. Ο κύριο Δημεσμάκη μου είχε δώσει υπόσχεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν 20 ε, χρόνια, ε, Πορτογαλός ε, ποιητής εδώ κινησε το φεστιβάλ του Σιροπάρλια και είπε στη γλώσσα μου μπορώ να ονειρευτώ τη θάλασσα. Θα μιλήσω πορτογαλικά λοιπόν. ο Homo sapiens ε, με συνεχή και προοδευτικό τρόπο και στη συνέχεια με επιταχυμένο τρόπο και στη συνέχεια με στιγμίο τρόπο τον 20ο αιώνα έγινε, στην, ε, μετατράπηκε στην κύρια μετασχηματιστική δύναμη της γεωλογίας του πλανήτη που μας ε, οδήγησε στο να μπούμε σε μια νέα γεωλογική εποχή, το ανθρωπόκαινο δεκάδες επιτυχημένης ανάπτυξη και βιομηχανική κοινοτομία μας έκαναν να ξεπεράσουμε τουλάχιστον τέσσερα από τα 9 όρια του πλανήτη. Οι θάλασσε και ωκεανοί που είναι στοιχεία σταθεροποιητικά για βιοκαιοφυσικών διαδικασιών και κυρίω ρυθμίζουν το κύκλο του άνθρακα σήμερα είναι αποδυναμωμένε τα προβλήματα πάνε πολύ πέρα από την υπερελίευση και από τη ρήπανση και τα χωροκατακτητικά είδη υποφέρουν και η οξύνηση, από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και πολλοί από αυτούς τους παράγοντες ελοπιδρούν με άλλους συνυπάρχοντες παράγοντες όπως η αύξηση του επίπεδου του νερού της θάλασσας, η απώλεια βιοπικιλότητας και η αύξηση περιοχών χωρίς οξυγόνο. Και πολλά από αυτά τα προβλήματα μπορεί να φαίνονται περιφερειακά και σίγουρα υπάρχουν τέτοια περιφερειακά ζητήματα. Το γεγονός είναι ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, από μια παγκόσμια σκοπιά. Ε, ο αντίκτυπο του ανθρώπου ε, πάνω στο θαλάσσιο συνστόσο του πλανήτη δεν έχει πολιτικά σύνορα. Οποιαδήποτε απάντηση είτε σε χώρια ύδατα είτε στην ανοιχτή θάλασσα θα πρέπει να γίνει από κοινέ πολιτικέ. Η παγκόσμια διακυβέρνηση και η τεχνική επιστημονική γνώση είναι οι πυλώνε για ένα βιώσιμο μέλλον. Χρειαζόμαστε συντονισμένα προγράμματα στις θαλάσσιες επιστήμες για να καταλάβουμε το ρόλο των ε, ωκεανών. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ένα στόχο marketing. πρέπει να είναι μια δέσμευση που θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να λάβει υπόψη τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξη μεταξύ περιοχών και χωρών. Ε, οι χώρε που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ε, για να έχουν χειρότερε περιβαλλοντικέ συνθήκε είναι οι λιγότερο αναπτυγμένε. Όμω αυτοί συνεισέφεραν λιγότερο στην κατάσταση του πλανήτη. Πρέπει να έχουμε προοδευτική και συνεχή η εστίαση στην παιδεία, στην κατάρτιση και στην έρευνα για να επιτρέψουμε ότι η νέα γενιά ε, των διαχειριστών των ωκεανών ε, ε, ασκούν τα δικαιώματά τους και τα καθήκοντά τους με μεγαλύτερη υπευθυνότητα για έναν υγιή ωκεανό. Ε, συνεχίζει να λειτουργεί το ρολόι και δεν έχουμε ωραίες ε, ατράκτους. Μπορούμε να καταλήξουμε σε γενοκτονία για ορισμένε περιοχές του ωκεανού και κατόπιν ε, για τον πολιτισμό μας. Στη συνέχεια ε, πρέπει ε, να έχουμε την ηθική ευθύνη μια γενιά ε, που κινητοποιείται. Σε ευχαριστώ αυτή τη νέα γενιά, αποτελεί ελπίδα. Thank Ευχαριστώ πολύ και που σεβαστήκατε και το χρόνο. Τώρα, η επόμενη ομιλήτρια είναι η Κλαούντια Μοντέριο Ντεαγκιάρ, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών. Έχετε τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους παρόντες και τους επιτρόπους και δεν μπορώ παρά να κλέψω κάποια δευτερόλεπτα από τα τρία λεπτά για να απευθυνθώ και να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ για όλη τη δέσμευσή της και το έργο της ε, για το γαλάζιο κόσμο, για τον κόσμο των θαλασσών και των ωκεανών. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σερό Σέντος, ε, παρά τις πολιτικές διαφορές που προσχωρίζουν. Είναι ένας ε, Πορτογάλος, ο οποίος χάραξε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο στον τομέα της θάλασσας και κατόπιν πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι ωκεανοί καθώς ε, βρίσκονται ε, σε προτεραιότητα του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίω ε, για να το προωθήσουμε στις επόμενες ευρωεκλογέ. Πρέπει να δείξουμε ότι ανησυχούμε για την κατάσταση αυτή, ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν αποδείξει ότι θέλουν να δράσουν απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται και επίσης να ε, απαριθμίσουμε όλους τους ακτιβιστές που αναφέρθηκαν εδώ. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, τον David Attenborough το, με το πρόγραμμά του στο BBC ε, ευαισθητοποιεί για να εργαστούμε περισσότερο για αυτή την προβληματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των πλαστικών στους ωκεανούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες προκλήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να προτείνουμε στρατηγικές ε, προσερμογής, μακροπρόθεσμες για την καταπολέμηση των επορριμμάτων αλλά και την κλιματική αλλαγή. Δύο δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ε, δαπανούμε για τι θαλάσσιε έρευνε, προωθώντας νέε υπηρεσίες και νέα προϊόντα για τη γαλάζια οικονομία. Ε, Παρ' αυτά χρειάζεται περισσότερες επιστημονικές γνώσεις και στοιχεία που να αναλύουν περισσότερο το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Ευρώπης ε, ε, θα παρέμβει στους ωκεανούς και θέλουμε να πεμπλοκάρουμε το δυναμικό των θαλασσών. Αυτό μπορεί να είναι το κλειδί για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Όλοι χρειαζόμαστε, είμαστε απαραίτητοι για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις πρέπει να συνεχίσουμε, όπως κάναμε και στην Επιτροπή Μεταφορών, σε μια γνωμοδότησή μας, εκφράζεται αυτό, να συνεχίσουμε τη στρατηγική για να ε, υπερασπίσουμε την περαιτέρω χρήση του γραπημένου φυσικού αερίου, αλλά και να αντικαταστήσουμε ε, τις πηγές ενέργειας που ρηπαίνουν περισσότερο. Θα πρέπει να έχουμε πιο διατομικές προσεγγίσεις και να ε, επικεντρωνόμαστε στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Επίσης, σε αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, θα πρέπει να εστιάσουμε και να αναφερθώ και στις άκρως απομακρυσμένες περιοχές ε, δεδομένου στις τοποθεσίες τους στον Ατλαντικό και στον Ινδικό κενό είναι θεμελιώδης για την μελέτη και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, του αντικτύπου στα θελασσικοσυστήματα οικοσυστήματα και στη βιοπικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να πω ότι θα προτείνω ένα κέντρο καταπολέμησης της θαλάσσιας ρήπανσης σε αυτές τις άκρως απορριμματισμένες περιοχές πιθανότητα στη είναι να ιδρυθεί για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να υιοθετήσουμε τρόπους καταπολέμησης της απειλής και αυτό ε, φυσικά σε συνεργασία με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα που βρίσκεται στην Πορτογαλία. Θα ήθελα να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στους νέους που είναι παρόντες εδώ. Όλοι να δεσμευτούμε για την καταπολέμηση της, των θαλάσσιων απεριμάτων, αλλά να αγωνιστούμε και για το μέλλον μας, να έχουμε κάθε φορά καλύτερες θάλασσες και ωκεανούς. Σας ευχαριστώ. Well, thank you. Thank you indeed, colleagues. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. We'll now listen to the contribution of... ε, θα ακούσουμε τώρα ε, ενδιαφερομένους και ενεχομένους φορείς. Παρακαλώ να συστηθείτε. Uh, ε, Mr. Thiago Pita Acuna, Chief Executive... Ε, το Διευθύνοντα Σύμβουλα ε, της ε, ε, του Ιδρύματος για τον ε, Γαλάζιο Ωκεανό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, Επίτροπε Βέλα, ε, πρώην μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, το σύστημα των ωκεανών είναι το πιο ευαίσθητο και ευπαθές του πλανήτη. Όμως, ο η δυνατότητά του να παράγει βιομάζα, να διατηρήσει τη βιοπικιλότητα ή να παράγει οξυγόνο υποβαθμίζεται ε, διαρκώς. Ως ε, συνέπεια, ο ωκεανός τελικά αλλάζει και ως προς τη βιοχημική του ε, σύνθεση. Αυτό πιέζει τον ωκεανό σε μια βαθιά και τον οδηγεί σε μια βαθιά περιβαλλοντική κρίση, η οποία δεν γίνεται πλέον αρκετά κατανοητή ε, και δεν έχει γίνει ακόμα αρκετά κατανοητή από τον άνθρωπο. Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει προσφέρει αρκετέ ε, λύσει για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα αυτό. Το 2020 θα είναι ορόσημο, χρονιά ορόσημο όχι για την επιτυχία μα, αλλά για τον οργανισμό των ωκεανών που εκπροσωπώ φόβου. Μπορεί να είναι και ορόσημο δυσαρέσκεια για την έλλειψη εξέβρεση λύσεων. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι πιο ισχυρά μεταξύ των νέων και είναι σαφή ενδείξεις της του. τους. Ε, το είδαμε και από τι παρεμβάσει των εκπροσώπων τους ε, προηγουμένω. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λάβουμε δράση. Ο ΙΕ αυτή τη στιγμή συζητά αυτού της ε, νέας συνόδου που θέλουν να διοργανώσουν Πορτογαλία και η Κένια για το μέλλον των ωκεανών. Ευχάριστες ειδήσει, αλλά δεν είναι το τελευταίο βήμα που μπορούμε να κάνουμε, ε, διότι με την εφαρμογή του στόχου της χιλιετία 14 ε, δεν θα λυθούν τα προβλήματα των ωκεανών. Πρέπει να βρούμε τα κομμάτια του πάζλ και, να... και τη συνολική εικόνα, τη διασύνδεση των κλιματικών αλλαγών με το τι γίνεται στους ωκεανούς ή το μοντέλο οικονομικής μας ανάπτυξης που εξαρτάται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στον πλανήτη και τον ανητικό αντίκτυπο που έχει αυτό το μοντέλο για τους ωκεανούς. Η διεθνή κοινότητα που εκπροσωπείται από τα μέλη του ΟΗΕ μεταξύ άλλων μπορεί να εγκρίνει στην επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για τους ωκεανούς μια σχετική συμφωνία, αλλά έχει σοβαρές ευθύνες και κοινωνία των πολιτών. Η ευθύνη αυτή είναι κάτι που συναισθανόμαστε πλήρως και ο οργανισμός μας προσπαθεί να σώσει ό,τι απομένει στους ωκεανούς, προσπαθώντας να προωθήσει νέες προστατευόμενες περιοχές με βιώσιμες αλληλευτικές ε, δραστηριότητες και ενισχύοντας μια γαλάζια οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρόμαστε που μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι η Περιφερειακή Κυβέρνηση των Αζωρών σε συνεργασία, σε εταιρική σχέση με, την, ε, με το Ίδρυμα ΟΕΤ και την, ε, τον δικό μας οργανισμό πριν δύο μήνες αποφάσισε να αφήσει ε, σε ανάπαυση ένα μεγάλο μέρος τη θαλάσσια ζώνη των, Αζωρών και να γίνουν αυτέ προστατευόμενε περιοχέ είναι ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής θαλάσσιας έκτασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που εκπροσωπεί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Πορτογαλία. Είναι τολμηρή και σημαντική απόφαση των Αζωρών, όχι μόνο για το δικό τους το αρχιπέλαγος ή για την Πορτογαλία μόνον, αλλά για ολόκληρο τον βόρειο ε, δυτικό Ατλαντικό ωκεανό, τον βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό. Ο οργανισμός των γαλάζιων ωκεανών δεν πιστεύει ότι θα πετύχουμε να έχουμε και ωκεανού μόνο με την διαφύλαξή του. Και η οικονομία μα είναι θέμα. Η δική μα οικονομική ανάπτυξη και το μοντέλο που έχουμε καθορίσει φαίνεται ότι δεν είναι συμβατό με την ε, βιωσιμότητα του πλανήτη. Υπάρχει σοβαρότατη επίγουσα ανάγκη να αλλάξει το μοντέλο αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τη φύση με άλλα μάτια. Είναι ένα κεφάλαιο ένα κεφάλαιο φυσικό και στο οποίο βασίζεται η ύπαρξη της κοινωνίας μας. Εάν γίνει κεφάλαιο η φύση, τότε οι δράσεις για να σώσουμε την φύση θα μπορούσε να θεωρηθεί οικονομική κίνηση. Είναι κεφαλαιακή επένδυση, όχι κόστος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το φυσικό κεφάλαιο να θεωρηθεί ως αντικείμενο που θα μπορούσε να το διαχειριστεί μια τράπεζα. Όπως είπε και η κυρία Δαμανάκη με το γαλάζιο ομόλογο ή με τη βιομάζα ε, που, με τις νέες προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχές. Κάτι που θα μπορούσε να το υπολογίσει στην τραπεζική του αξία Παγκόσμια Τράπεζα. Παρομοίως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυχώς στην ενεργειακή της πολιτική πρότεινε μέτρα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για μια ατζέντα για τους ωκεανού που να προωθεί την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των ωκεανών. Κυρίες και κύριοι, ε, όσο αναβάλουμε ε, την δράση, τόσο πιο ριζοσπαστικές αλλαγές θα χρειαστούν. Οι νέες γενιές δείχνουν ότι δεν έχουν άλλη υπομονή. Ε, ο θυμός θα φουντώσει εάν οι θύνοντες παγκοσμίως δεν λάβουν αν δεν αναλάβουν ευθύνες και δεν αναλάβουν μέτρα για τις θαλάσσιες περιοχές και τα διάφορα αρπακτικά ή τα κοράλια ή ε, για όλα τα είδη που ζουν στη θάλασσα. Πρέπει να σταματήσουμε την περιβαλλοντική υποβάθμιση και να σταματήσει ο φαύλο κύκλο όπου η περιβαλλοντική υποβάθμιση θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική ύφεση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Ο Δόκτωρ ε, Βλάντιμιρ ε, Ριαμπίνιν, εκτελεστικός γραμματέας της ε, διακυβερνητικής οκενογραφικής επιτροπής και αναπληρωτής γενικός ε, διευθυντής της UNESCO. Για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω να σας χαιρετήσω εξ ονόματος της κυρίας Όντρια Ζουλέ, ε, Διευθυντού της UNESCO. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Υπάρχει μια διάσταση παγκόσμια εδώ, διάσταση των Ηνωμένων Εθνών και θέλω να μιλήσω για το ρόλο της ωκεανογραφίας και της επιστήμης των ωκεανών για το μέλλον. Θέλω να απευθυνθώ στους νόους και να σας πω ότι είναι πραγματικά πολύ σπουδαία επιστήμη αυτή και επάγγελμα και θα βρείτε και δουλειά ε, ε, στον 21ο αιώνα να ασχοληθείτε με αυτά τα θέματα της ε, ωκεανογραφίας. Η Επιτροπή μας έχει ένα ρόλο καθοδήγησης ε, της επιστήμης για τους ωκεανούς από πλευράς ΟΗΕ. Παγκοσμίω. Η Ευρώπη όμως, είναι ο υπαριθμόν ένα ηγέτης στην επιστήμη. Είναι τρία τα κέντρα ε, τα ισχυρά. Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και ε, Δυτικός Ειρηνικός. Συνεργαζόμαστε πολύ παραγωγικά και γόνιμα με την Ευρώπη Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης. Ε, υπάρχουν βάσεις δεδομένων στην Ευρώπη, όπως είναι η Emotnet. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, για τον ειδικό σχεδιασμό για τη θάλασσα, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι το 1 τρίτο των ΑΟΣ παγκοσμίω μέχρι το 2030 να καλύπτεται από εγκεκριμένες από τις κυβερνήσεις ε, προσπάθειες, δράσεις και σχέδια, ειδικά για τη θάλασσα. Συνεργαζόμαστε και με τη Γενική Διεύθυνση Επιστήμης και Έρευνας ε, και ε, θα συνεισφέρει πολύ το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη, Horizon Europe, αλλά και πολλά υποσχόμενα είναι και τα παρατηρητήρια. Πού βρίσκονται επιστήμες των ωκεανών, η ωκεανογραφία. Ε, έχουμε μια πρόσφατη ανάλυση που λέει το εξής. Είναι αρκετά καλή επιστήμη για να φωτίζει ε, την κατάσταση. Ξέρουμε πόσο διοξείδιο του άνθρακα απορροφάει ο ωκεανός, πόσο θερμότητα απορροφά ο ωκεανός, τι γίνεται με το οξυγόνο, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε καλές λύσεις. Η κατάσταση μας θυμίζει τα όσα συνέβησαν και για το κλίμα το 2008. Υπήρξε η επιστήμη και τα στοιχεία, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία για δράση και ούτε δράση υπήρχε. Και τώρα θα πρέπει να δράσουμε πραγματικά για να μπορέσει η επιστήμη να είναι αποτελεσματική. Η Επιτροπή μας ε, ε, έκανε προτάσεις ε, στον ΟΗΕ ε, για τις επιστήμες των ωκεανών που να προτείνουν λύσεις όμως προσανατολισμένες ε, στην ε, πράξη. Και πραγματικά συμμετέχουν πολλοί και ο κύριος Σάντος. Να σας πω ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι σε διάφορους τομείς να έχουμε ρηξικέλευθες δράσεις, χαρτογράφηση, παρατήρηση, δεδομένα, κατανόηση των οικοσυστημάτων και των μεγάλων βαθών τη δυνατότητα οικοδόμησης ικανοτήτων. Καταλαβαίνετε ε, πώς ε, έτσι αυξάνονται οι γνώσεις μας για τον ωκεανό ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι τομές. Είναι πολύ σημαντικά, καλά σχεδιασμένα και θα μπορέσουμε σε πολλούς τομείς να έχουμε ουσιαστικά ωφέλη. Διαχείριση παρακτήων ακτών, ε, προσαρμογή και μετρίαση του, της κλιματικής αλλαγής, ε, χωροταξικός σχεδιασμός στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι τομείς δραστηριοτήτων ε, που μας οδηγούν να κάνουμε τους ωκεανούς παραγωγικούς, αποδοτικούς, με μια γαλάζια οικονομία και όχι ε, εις βάρος της υγείας των ωκεανών. Ακριβώς αυτή είναι η ιδέα της ωκεανογραφίας, της επιστήμης των ωκεανών και προσεχώς θα έχουμε μια παγκόσμια ε, διάσκεψη στην Κοπενχάγη το Μάιο. Αναφέρθηκε και ο Τιάγκο προηγουμένως ε, μια διάσκεψη για τις δράσεις που απορρέουν από την επιστήμη και τα δεδομένα. Ελπίζω πάρα πολύ η Ευρώπη να ε, στερνιστεί αυτό το μήνυμα και να βοηθήσει στην ωκεανογραφία και έχουμε για αυτή τη δεκαετία και έχουμε και ένα σλόγγαν «Ο ωκεανός που χρειαζόμαστε ε, για το μέλλον ε, που θέλουμε». Τώρα μιλάμε για την επιστήμη που χρειαζόμαστε για τον ωκεανό που θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα τόσα μας είπατε. Και τέλος ε, θα δώσω το λόγο στον Πίτερ Χέρτσικ, είναι εκτελεστικός διευθυντής ε, στο κέντρο GMR ε, στο Κίελο, στη Γερμανία. Για την έρευνα σοκενούς, πέρα παρακαλώ, έχετε το λόγο. Να σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τους καθαρούς ωκεανούς και θάλασσες από τη σκοπιά της έρευνας και θα ξεκινήσω με το 70%. Το ακούσατε πολλές φορές σήμερα. Το 70% καλύπτεται από ε, τους ωκεανούς, έχουμε την, ε, διάφορους ωκεανούς, την Αυξηνοπόντο, τη Βαλτική, τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Θάλασσα, τον Ειδικό Κενό, τον Ατλαντικό, τον Ελληνικό. Και το 70% λοιπόν του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό ε, από των ωκεανών και γι' αυτό ζούμε σε ένα γαλάζιο πλανήτη. Είναι λοιπόν σημαντική η ωκεανή για μας, όχι μόνο ε, λόγω των μεγεθών τους, αλλά γιατί είναι ένα μεγάλο οικοσύστημα στον πλανήτη. Και έχουμε ακούσει και πάλι ότι υπάρχει πρόβλημα με το οξυγόνο. Παρέχει λοιπόν ο ωκεανός το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε και αυτό οφείλεται στη δραστηριότητα των μικροοργανισμών στον ωκεανό. Αν ε, δεν μας κάνουν αυτή τη χάρη δεν θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, δεν θα ήμασταν εδώ σε αυτή την αίθουσα. Αυτό αποτελεί λοιπόν σημαντική λειτουργία και υπηρεσία των ωκεανών. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν, μάλλον απορροφούν το 30% των του άνθρακα από την αρχή της βιομηχανικής εποχής και το 30% σημαίνει ότι δεν θα μιλούσαμε σήμερα για το στόχο 1,5-2% ενώ θα ήμασταν σε μια πραγματικότητα 4-5 βαθμών Κελσίου. Μας έχει κάνει μεγάλη χάρη λοιπόν ο Γκένος και πάλι εδώ, αλλά ε, ξέρετε... Ε, το ότι απορροφάτε το διοξείδιο του άνθρακα του ε, ουσιαστικά έχει και ένα τίμημα, προκαλεί τοξίνηση. Επίσης ε, και και ωκεανός ε, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θερμότητας που παράγουμε και επίσης παρέχει τροφή για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι λοιπόν οι ωκεανοί είναι ζωτικοί για μας, το ακούσαμε και στο παρελθόν. Ο ωκεανός ε, ουσιαστικά αποτελεί το σύστημα στήριξης ζωή του πλανήτη. Ε, πρόκειται για έναν ασθενή όμως την εντατική. Αλλά δεν είμαστε καλοί γιατροί, δεν προσέχουμε τους ωκεανούς μας, ε, γιατί ε, εδώ με την πίεση που βάλουμε στους ωκεανούς προκαλούμε οξύνηση στους ωκεανούς και φερούμε το οξυγόνο. Αυξάνονται οι περιοχές που έχουν το οξυγόνο σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Αυξήνουμε την θερμότητα των ωκεανών, ρηπαίνουμε τους ωκεανούς, τα πλαστικά. Ε, είναι ένας παράγοντας χημικής, αλλά έχουμε και χημικού τύπου ρήπανση, βιολογικού τύπου ρήπανση. Επίσης, ε, ζημιώνουμε την βιοπικιλότητα των ωκεανών. Δεν έχουμε καν ανακαλύψει όλη τη βιοπικιλότητα, αλλά έχουμε προκαλέσει βλάβη σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτή. Αναφέρθηκε και η υπεραλίευση και το θέμα των χωροκατοκτητικών ειδών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε σήμερα, όμως υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα που ανακύπτει το 2050 θα έχουμε 50% περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη, δηλαδή 10 με 10,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι το 50% περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 50% περισσότερα τρόφιμα, περισσότερη ενέργεια και 50% περισσότερους πόρους. Και κάποια θα πρέπει να έρθουν από τους ωκεανούς. Κάποια από αυτά. Έτσι λοιπόν η πίεση στους ωκεανούς αυξάνεται ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα γη ωκεανό για υγιεί ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό απαιτεί περισσότερη έρευνα που να προσανατολίζεται στη λύση. Η βασική έρευνα αποτελεί τη βάση, αλλά χρειαζόμαστε έρευνα που να προσανατολίζεται σε λύση, μεγαλύτερο συντονισμό τη έρευνα και πιο στοχευμένη χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να τάσουμε σε προϊόντα και δράσει. Η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα τη σωτηρία των ωκεανών μας για τις επόμενες γενιές στον πλανήτη. Νομίζω ότι αυτό έχει αναφερθεί και στο παρελθόν και θα ήθελα να είμαι κάπως πιο κλητικός στο σημείο αυτό γιατί πάντοτε αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τους ωκεανούς καθώς αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα και αφιερώσαμε όλο το απόγευμα σήμερα στη συζήτησή του, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ίσως λοιπόν θα χρειάζεται περισσότερη προβολή, περισσότερη ηγετική στάση και δράση από την ευρωπαϊκή πλευρά όταν ε, μιλάμε για τη διάσωση των ωκεανών μας και των θαλασσών μας. Σας ευχαριστώ. Well, Ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε στο τέλος του πάνελ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας που προσπάθησαν να μας δώσουν μια συνολική εικόνα του τι είναι το διακύβευμα τι μπορούμε να κάνουμε για τη διαφύλαξη των ωκεανών μας, πόσο σοβαρά παίρνουμε το θέμα αυτό και ότι παρά όλα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρονική πίεση. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να προσκαλέσω τον συνάδελφο Χένκελ που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, για την ε, Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια, να αναλάβει το επόμενο πάνελ για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. All over Europe, people are getting ready to vote in the European elections in May. Whoever you are, wherever you are, you can get involved